Επεξηγήσει eh, eh. Επεξηγήσεις ψήφου λοιπόν τώρα. Ξεκινάμε με την έκθεση Μπέρες όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού 1927. Έχω τρεις ομιλητές. Γιάρ, είναι ο πρώτος ομιλητής. Παρακαλώ. Θα ήθελα στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από πλευράς μας να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατηρήση είναι είμαι πραγματικά ενθουσιώδης υποστηρικτή του Ευρωπαϊκού Ταμείου αυτού, διότι εξυπηρετεί απλά όταν έχουμε προβλήματα στην προσαρμογή στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία μπορούμε να βοηθήσουμε με τα κονδύλια αυτού του Ταμείου και μπορούμε να διατηρήσουμε την πίστη στην παγκοσμιοποίηση στους ανθρώπους λέγοντας ότι τα μειονεκτήματα που δημιουργούνται από την παγκοσμιοποίηση αντισταθμίζονται με αυτές τις δράσεις, με αυτά τα κονδύλια. Από την άλλη πλευρά ανήκω και στους σκεπτικιστές που λένε ότι γι' αυτό το Ταμείο πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένος τίτλος δημοσιονομικά διότι πιστεύω ότι δεν μπορεί κανείς να να προγραμματίζει καταστροφές και υπάρχει ο κίνδυνος ε, όταν δεν έχουν εξαντληθεί κονδύλια μετά να μοιράζονται κονδύλια και ουσιαστικά δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι καταστροφή με αυτόν τον τρόπο. Είμαι υπέρ, αλλά πρέπει να υπάρχει και επιφύλαξη και σύνεση στο σωστό βαθμό. Αυτό είναι το σωστό. Ευχαριστώ πρώτα. Ευχαριστώ θερμά. Αγαπητοί συνάδελφοι, Όσοι από εσά δεν θέλετε να υποβάλλετε επεξήγηση ψήφου, παρακαλώ να καταλήψετε το εμικύκλιο για να συνεχίσουμε εμεί. Ο κύριος Σάναν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, έτσι τελειώνει τελικά το πράγμα. Αντιμετωπίζουμε την κρίση χρησιμοποιώντας ένα απίστευτο ποσό, 3-3 ευρώ το μυαλό μας δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί τέτοια ποσά. Οπότε απορρέουν δύο ερωτήματα εδώ. Ποιος ε, θα μας ε, τα εγγυθεί αυτά. Τελικά πρόκειται για ένα δάνειο το οποίο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα πρέπει να το καλύψει, να το εγγυθεί. Από την άλλη μεριά αγοράζει ομόλογα τα οποία δεν έχουν πια καμία απολύτως αξία στην ε, αγορά. Θεωρούνται junk. Τελικά μήπως ο φορολογούμενος. Δεύτερον, και από ποιον. Ποιος έχει δηλαδή τα τρία 3 Αν κάποιος ειχε τρία 3-3, κάπου θα τα είχε ήδη χρησιμοποιήσει. Οπότε τελικά εμεί δανειζόμαστε από τις επόμενες γενιές. Αυτό κάνουμε. Και όπως έλεγε και όπως λένε έχουμε ακούσει, τελικά όλα αυτά θα πλήξουν τις επόμενες γενιές και δεν θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο και να την πληρώσουν τα παιδιά μας. Ευχαριστούμε κύριε Ανάν. Ο κύριος Κέλλη. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, τώρα στον αφορά την έκθεση αυτή για το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης, ε, α, α, γι' αυτό συζητάμε. Το... Ή το επόμενο. Yeah. Κύριε Κέλλη, επεξήγηση ψήφων για την έκθεση κυρίας Μπερές. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Μπερές, λοιπόν. Να το κάνουμε τώρα, μιλήσω τώρα, μπορώ να μιλήσω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η σημασία είναι διπλή. Πρώτα απ' όλα δίνεται βοήθεια πραγματική στους ανέργους για να βρουν ταχύτερο δυνατόν δουλειά. Σε άλλο επίπεδο δίνει θάρρος σε εκείνους που είναι πολύ πικραμένοι, στραχωρημένοι, δεν είναι άνεργοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το είδα στην Dell, στην Waterford Crystal και στην Tok Tok. Ε, υπάρχουν κάποιοι που είναι πρόθυμοι και θέλουν να βοηθήσουν τους εργαζομένους. Υπάρχουν προβλήματα με το Ταμείο. Υπάρχουν τροπολογίες τώρα και άλλες αλλαγές θα χρειαστούν μετά το 2013, γιατί αυτό το Ταμείο θα χρειαστεί επιμακρών, δυστυχώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Άλλος ο οποίος θέλει να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο ψήφισε. Όσον αφορά την έκθεση της κυρίας Μπερές, δεν υπάρχει άλλος που θέλει να κάνει επεξήγηση ψήφου. Επεξήγηση ψήφου για την κατάσταση στην Παλαιστίνη τώρα. Ο κύριος Ταραντ έχει το λόγο. Ο κύριος Ταραντ απουσιάζει. Ο κύριος Τακούλα λοιπόν έχει το λόγο. πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω σε σχέση με αυτό το εξή ε, για αυτή την ψηφοφορία. Συχνά έχουμε ψηφοφορίες ε, που αφορούν τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές και περί αυτού πρόκειται και σε αυτή την ψηφοφορία εξίσου. Πολλοί επανειλημμένα κάνουν λόγο για δημοκρατία, ελευθερία της έκφρασης, θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιώματα του ανθρώπου κτλ. Γνωρίζουμε όμως όλοι ότι το Ισραήλ είναι η μόνη δημοκρατική χώρα σε αυτή την περιοχή της Μέσης Ανατολής και γι' αυτό αξίζει, θα έπρεπε να αξίζει πραγματικά υποστήριξη από πλευρά μας. Ως προς όλα αυτά είναι θλιβερό το ότι αυτό το μήνυμα αποστάθηκε από την πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου όπως έγινε. Όμως παρόλα αυτά βλέπω ότι πολλοί στη δική μου την πλευρά καταψήφισαν αυτό το ψήφισμα και που βρίσκονται στο πλευρό του Ισραήλ ως σύμμαχοι, ως ε, υποστηρικτές και θέλουν να μεριμνήσουν ώστε η Ιερουσαλήμ να εξακολουθεί να είναι η πρωτεύουσα, η ε, πόλη του ε, κράτους αυτού και θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει και σε σχέση με τους, ε, τα γειτονικά κράτη θα πρέπει να μπορέσει να αντανακλάται εκεί η δημοκρατία. Ε, Πρόεδρε, πιστεύω εγώ ότι οι περισσότεροι ευρωβουλευτές ε, στο Ευρωπαϊκό μας Κοινοβούλιο σε αυτό το θέμα βρίσκονται διάμεσα, δηλαδή στο πλευρό των ανθρώπων των πολιτών. Μπορεί τώρα να έχει κανείς αντιπαράθεση λέγοντας αν οι Παλαιστίνοι θα πρέπει να ενταχθούν στο, στον Οργανισμό Ηνωμένων ως ανεξάρτητο κράτος ή όχι. Από την άλλη όμως πλευρά κατανοώ και τις ανησυχίες που υπάρχουν μετά από τόσες δεκαετίες να μην έχουν υπάρξει χειροπιαστά αυτά αποτελέσματα και θα πρέπει να προχωρήσουν τα μέτρα ε, οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ποτέ δεν μπορούν να είναι μονομερή αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πρέπει να είναι αμφωτέρωθεν και αναμένουμε σαφή μηνύματα από το ίδιο το Ισραήλ και θα πρέπει για το δεύτερο, για την πολιτική δηλαδή των επικισμών από το Ισραήλ να την λάβουμε σοβαρά υπόψη. Δεν είναι καθόλου επικοδομητική και ούτε οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση. Ο κύριος Ρέπο είναι επόμενος. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε η διαδικασία, η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή πρέπει να μπορέσει να συνεχιστεί και να σταθεροποιηθεί όπως λέμε σε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος. Το δικαίωμα αυτοδιάθεσης και ε, αυτοπροσδιορισμού των Παλαιστινίων και το δικαίωμα του Ισραήλ να έχει ένα ανεξάρτητο ασφαλές κράτος σε ασφαλή σύνορα θα πρέπει να διασφαλίζεται οπωσδήποτε. Η απογοήτευση του Προέδρου Αμπά είναι κάτι το απόλυτα κατανοητό. 20 χρόνια διαπραγματεύσεις είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως στην διεθνή πολιτική πολιτική πρέπει να λάβουμε υπόψη και την αλληλουχία των πραγμάτων, χρονικά την αλληλοδιαδοχή τους. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ομιλεί με μια ενωμένη φωνή. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια ενιαία θέση όσον αφορά την αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή και θα συνεισφέρουμε για την εξέβρεση μια ειρηνική λύση. Η μόνη δυνατότητα μακροπρόθεσμα ειρήνη σε αυτή την περιοχή περνά μόνο μέσα από τον πολιτικό διάλογο και τι διαπραγματεύσει. Οι εταίροι στι διαπραγματεύσει πρέπει να καταλήξουν σε, ένα, σε μια στρογγυλή τράπεζα και να διαπραγματευτούν επιτέλους. Και άσχετα από το τι θα γίνει από τη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις. Η κυρία Εσάγη έχει το λόγο. Εγώ σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να δώσω μια επεξήγηση ψήφου για την, το ψήφισμα για την Παλαιστίνη, διότι η δική μου θέση θα έπρεπε και αυτή να καταχωρηθεί στα πρακτικά. Υποστηρίζω αυτό το ψήφισμα πρέπει να πω. Δεν, μπορώ να υποστηρίξω αυτό το ψήφισμα, δεν μπορώ ούτε το ψήφισμα ούτε το περιεχόμενό του διορθώνεται να υποστηρίξω. Διότι είναι σημαντικό να υπάρξουν δυνατότητες διαπραγμάτευσης ε, από τους εταίρους γύρω από μια τράπεζα διαπραγματεύσεων. Σημαντικό όμω είναι επίσης η κατάσταση όσον αφορά την Ιερουσαλήμ να αποσαφινιστεί και τα σύνορα να προσδιοριστούν με σαφήνεια. Η ιδέα εμπιστοσύνη και των δύο πλευρών πρέπει να είναι αναγκαία προϋπόθεση. Αυτή όμως η προϋπόθεση δεν μπορεί να επιβληθεί έξωθεν εκ των έξω. Πρέπει και οι δύο πλευρές να καλλιεργήσουν το κλίμα εμπιστοσύνη ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν υποστηρίξει το κράτος των Παλαιστινίων τότε σίγουρα αυτό θα είναι μια πολύ δύσκολη θέση που θα δημιουργηθεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα μπορέσουμε να την ε, υπερασπιστούμε. Ευχαριστώ. Mr. President. Ο Μπάνερμαν. Είμαι υπέρ του Ισραήλ, αλλά είμαι και επικριτικός φίλος του Ισραήλ. Εγώ ο ίδιος έχω δουλέψει στην διαδικασία την ειρηνευτική στη Βόρεια Ιρλανδία εκ μέρου τη Βρετανική κυβέρνηση. Εννοείται ότι δεν μπορεί να λυθεί με στρατιωτικό τρόπο το ζήτημα, αλλά πολιτικά. Και οι νομικοί αυτοί διακανονισμοί δεν βοηθούν τη διαδικασία. Ξέρω ότι υπάρχει κακή μεταχείριση, ξέρω ότι χρειαζόμαστε ένα κράτος που να ζει ειρηνικά δίπλα στο Ισραήλ. Όμως δεν είμαι σίγουρος ότι το μέτρο αυτό που μπορεί να είναι καλή διαπραγματευτική τακτική μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία του κράτους της Παλαιστίνης. Δεν νομίζω ότι είναι ο σωστός τρόπος, γι' αυτό και κράτησα θέση αποχής. Πάντως, επιθυμώ η ειρηνευτική διαδικασία να προχωρήσει. Νομίζω ότι αυτό είναι ζωτική σημασία. Και μόνο οι διαπραγματεύσει, όπω το είδαμε και στην Βόρεια Ιρλανδία, μόνο αυτέ μπορούν να οδηγήσουν σε μια πολιτική λύση από την οποία έχουν αποφεληθούν όλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κάμπελ Πάνερμαν. Άλλο κανεί για το ψήφισμα όσον αφορά την Παλαιστίνη. Όχι. Συνεχίζουμε λοιπόν και περνάμε τώρα στο Ρίο συν 20, τη διάσκεψη κορυφή. Παρακαλώ κύριε Πασέσκου να μας εξηγήσετε πώ ψηφίσατε. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρόεδρε, πιστεύω ότι οι εξελίξεις και μια πράσινη οικονομία αποτελεί την εναλλακτική λύση της εκμετάλλευσης ορυκτών. Εγώ καταψήφισα την παράγραφο 46 του ψηφίσματος γιατί η εφαρμογή της μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικά προβλήματα εφόσον θα αυξηθεί η τιμή του ηλεκτρισμού για τον τελικό καταναλωτή. Η ε, έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα που επηρεάζει βέβαια τα πράγματα έχει κάποιες οικολογικές επιπτώσεις. Εμείς θέλουμε την βιοπικιλότητα και πάντα συμμετείχαμε στην εκπόνηση διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. Η Ρουμανία το στηρίζει αυτό, στηρίζει και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Αλλά δεν θέλω να σταματήσει η πυρηνική ενέργεια και να μην χρησιμοποιείται πια στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μίξ, γιατί είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και συγχρόνως είναι και μία μη ακριβή ενέργεια. Πρέπει να, το να σταματήσουμε να φτιάχνουμε νέους πυρηνικούς σταθμούς δεν είναι κάτι από το οποίο έχει να αποφεληθεί το περιβάλλον. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρέπο έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, για το ε, ψήφισμα αυτό όσον αφορά τον πλανήτη Ρίο Συνήκωση, ίσω θα μπορούσε να υπήρχε μια κοινή κατευθυντήρια γραμμή. Ένα από τους βασικού στόχου είναι να διασφαλίσουμε μια πρόσβαση που να προστατεύει τους πόρους της γης και για τη σημερινή γενιά και για τις επόμενες. Μόνο έτσι θα έχουμε αηφόρο ανάπτυξη και μόνο έτσι θα μειωθεί η ένδυα στον κόσμο. Εγώ θα ήθελα το ΡΙΟ να προωθεί μια αηφόρο ανάπτυξη και να βρεθεί μια λύση για μια πιο πράσινη οικονομία και για μια πιο πράσινη ενέργεια. Επιπλέον πρέπει να, να δούμε με ποιο τρόπο θα έχουμε μια πιο κοινωνική ε, κοινωνία και πόσο θα υπάρχει περισσότερη δικαιοσύνη σε αυτήν. Μία αηφόρος και πράσινη κοινωνία σημαίνει ότι σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα, την πολιτιστική πολυμορφία, τη θρησκευτική πολυμορφία και ότι φροντίζουμε να υπάρχει και ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που είχα τη δυνατότητα να υποστηρίξω αυτή την έκθεση. Υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα που τίθενται. Θα αναφερθώ σε τρία μόνο μόνος. Πρώτα απ' όλα θα εξασφαλίσουμε τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και θα πρέπει πάντα να παραμείνει δημόσια αγαθό και υποστηρίζω πλήρω την έκκληση αυτή, για δηλαδή το δικαίωμα στο νερό και στα, στην υγεία, στις υγειονομικές υπηρεσίε ε, πρέπει να καλύπτεται. Χρειάζεται και πρόσβαση στους, ε, στις θάλασσες για όλους τους, για στους πόρους, συγγνώμη, για τους ε, πληθυσμούς και για του γενετικά τροπημένου οργανισμού. Λοιπόν, ακάθαρε από όσου υπερκρατούν για του γενετικά τροπημένου οργανισμού, όλοι θα πρέπει να υποστηρίζουν την ασφαλή πρόσβαση στου σπόρου. Θα ήθελα να αναφερθώ στι παραγράφου 59 και 60, όπου περίπου 98% εκφράσαμε τι ανησυχίε που είχαμε όσον αφορά το, το, τα μέτρα για τα δάση που θα, ε, θα οδηγήσει σε αποψήλωση των δασών στον Αμαζόνιο. Και ο Επίτροπο, ο κ. Τεκούχτεν, το μεταξύ, εξακολουθεί να προχωρεί για να πετύχει συμφωνία Μερκοσούρ, συμπεριλαμβάνοντα και τις μεγάλες αγωγέ βοηθού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αποδάσωση του Αμαζονίου θα αυξήσει τα προβλήματα. Λοιπόν, διαφωνούν τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκφράζεται μια άποψη μια πλευρά και η άλλη πλευρά αγνοεί αυτές τις απόψεις. Ευχαριστώ κύριε Χάρκιν. Ο κύριος Κέλλη θέλει να πει κάτι, να πει μερικά λόγια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα παρακολούσα τη συζήτηση στο απόγευμα, ήθελα να είμαι στη συζήτηση στο απόγευμα, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα να συμμετάσχω. Το Ρίο ΣΥΝ 20 είναι σημαντικό θέμα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τον κόσμο πιθανότατα είναι τώρα πιο σοβαρά από ποτέ. Η αποψήλωση των δασών, από ε, περίμωση, υπερβολική αλίευση, ε, παροχή ε, καθαρού νερού, αλλαγή του κλίματος. Θα πρέπει έτσι σε παγκόσμιο επίπεδο να αντιμετωπιστούν. Δεν έχει νόημα να κάνει να παίρνει μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της και να βρίσκεται σε ισχυρή θέση ε, και να, βρίσκεται, να μπαίνει κόσμο στη φτώχεια και άλλοι να κάνουν τα δικά του. Τα παγκόσμια προβλήματα χρειάζονται παγκόσμιε λύσει, γενικέ λύσει και ελπίζω από αυτή τη σύνοδο να βγουν κάποια μέτρα. Όπω είπε χθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πολιτική σύμφωνα με την οποία πρώτα χρειαζόμαστε ανάπτυξη, μετά καθαρίζουμε, είναι κάτι απαράδεκτο. Είναι κάτι που δεν μπορεί να ισχύει και είναι απαράδεκτο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Η κυρία Μοκουλιένε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Υπερψήφισα αυτή την πρόταση ψηφίσματος που κατά το μάλλον ήταν αντανακλά μια ρεαλιστική προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αηφόρο ανάπτυξη. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ότι καταφέραμε να αποδυναμώσουμε τα όσα αναφέρονται στο εδάφιο 46 όσον αφορά την απαγόρευση για την δημιουργία νέων ε, πυρηνικών σταθμών. Τέτοιου είδους πράγματα δεν ε, ανταποκρίνονται στις απαιτήσει ε, των κρατών μελών και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό αν αποφασίσουμε να μην χρησιμοποιήσουμε την πυρηνική ενέργεια, αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ακόμα εξάρτηση από ενεργειακές πηγές. Τα ενεργειακά θέματα είναι θέματα των κρατών μελών και πρέπει να διασφαλίσουμε υψηλέ προδιαγραφέ, ακόμα και υψηλέ προδιαγραφέ για του πυρηνικού αντιδραστήρε. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πόρη και είναι επιτακτική ανάγκη να αναπτύξουμε αυτή τη συνιστόσα τη πυρηνική ενέργεια, όχι μόνο τώρα, σήμερα, αλλά και στο μέλλον. Και θέλουμε να υποστηρίξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν μάλλον αρνητικό όσον αφορά μη παραδοσιακές ενεργειακές πηγές. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάτεν Μάικε, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ από πλευράς μου υπερψήφισα αυτή την πρόταση ψηφίσματος και πρέπει να πω ότι η διάσκεψη του Ρίο μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο ως διάσκεψη. Μπορεί να δείξει ποιες είναι οι σωστές κατευθύνσεις, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε χειροπιαστά αυτά αποτελέσματα και σε προτάσεις που στη συνέχεια θα υλοποιηθούν και θα πάρουν σάρκα και οστά. Μόνο ωραίοι δεκάρικοι λόγοι και δηλώσεις ε, δεν επαρκούν. Έχουμε πια ε, πάρα πολλούς τέτοιους λόγους και ε, διακηρύξεις και δεν φτάνουν. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η εκπροσώπηση της από μη σε οργανώσεις να υιοθετήσουν μια κοινή θέση ως πλατφόρμα και να διαδραματίσουν ένα επικοδομητικό ρόλο όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να συναγάγουμε τα σωστά συμπεράσματα από τα μαθήματα του παρελθόντος και τα βιώματά μας. Και είδαμε, με άλλα λόγια, ότι πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο και τότε μπορούμε μόνο να προοδεύσουμε όταν από κοινού κινηθούμε όλοι προς μια κοινή κατεύθυνση και έχουμε επικοδομητική συνεργασία. Αυτό είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Άλλος για το Συνήκωση δεν θέλει άλλο το λόγο. Μπορούμε να αρχίσουμε με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, επεξηγήσει ψήφου. Η κυρία Χάρκιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω πλήρω αυτό το ψήφισμα και πιο συγκεκριμένα το αίτημα του Κοινοβουλίου, την έγκριση του Κοινοβουλίου να συνεχιστεί το Ταμείο αυτό πέρα από την παρούσα ισχύ είναι κάτι που είναι σαφέ μήνυμα από το Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε το Ταμείο και ότι έχει αξία αυτό το Ταμείο και σίγουρα ελπίζω το Συμβούλιο να ακούει προσεκτικά σε αυτά που λέμε. Ναι, πράγματι το ψήφισμα αναφέρει ότι θα πρέπει να κάνουμε αλλαγέ και μπορούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία του Ταμείου. Σίγουρα μπορούμε να βελτιώσουμε την έγκαιρη λειτουργία του και τους, να βελτίωση τη χρηματοδότηση. Εξασφαλίσουμε ότι το Ταμείο ανταποκρίνεται σωστά στι ανάγκε των εργαζομένων καθώ και ότι ασχολείται με τα προβλήματα τη κακή προσαρμογή των διαφόρων προσόντων. Σήμερα το πρωί κάποια θέματα όσον αφορά το να ε, ξεφύγουν από τι ευθύνε τους οι επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Ε, εάν το μελετήσει καλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σίγουρα μπορούμε να γίνουμε πιο αυστηροί, αλλά αυτό το χρησιμοποιούν τα μέλη κάποια φορά για δικαιολογία για να μην, ε, ε, χρησιμοποιήσουν το, να μην υποστηρίξουν το Ταμείο. Καλωσορίζουμε τον Εύρο, θα γίνει η, η επανεξέταση του πώς το τεγεμίου τον Νοέμβριο. Ε, από αυτά που εμπεριέχει η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ευπρόσδεκτα, και η πρόταση να χρησιμοποιηθούν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι γεωργοί στο ταμείο αυτό. Το καλωσορίζω. Ευχαριστώ, κυρία Χάρκιν. Κύριο Φάμον, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταψήφισα την έκθεση αυτή όσον αφορά το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, γιατί πιστεύω ότι είναι άχρηστο και θα έπρεπε να ακυρωθεί. Νομίζω ότι η βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν να κάνουν με την παγκοσμιοποίηση πρέπει να υπάρχει σε εθνικό επίπεδο και όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργεί ανισότητες, γιατί τελικά μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στα κονδύλια αυτά. Εξάλλου την ε, παγκοσμιοποίηση ε, την ε, αντιμετωπίζουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και απλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να αποφεληθούν από το ταμείο αυτό, γι' αυτό και με κατά. Τέλος, όσον αφορά τώρα την ε, συμφωνία εταιρική σχέση στον τομέα τη Αλία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μαρόκου. Παρακαλώ. Κύριε Ρεπό, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε να κάνουμε με μια κοινότητα αξιών η οποία βασίζεται στο γεγονός ότι θέλουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Συμφωνία εταιρική σχέση, λοιπόν, πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει εταιρικέ σχέσεις οι οποίε δεν ευθυγραμμίζονται με τις βασικές της αξίες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσο η συμφωνία αυτή θα είναι μια συμφωνία από την οποία θα αποφεληθεί ο κόσμος στη Δυτική Σαχάρα ή όχι. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε νομική πραγματογνωμοσύνη όσον αφορά αυτό το θέμα. Όσον αφορά τις εξωτερικές της σχέσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει η διένεξη στην, ε, με το Σαραούι να λήξει στη Δυτική Σαχάρα, δηλαδή όσο γίνεται καλύτερα. Ευχαριστούμε. Ρωμέβα Ιρουέβα. Για άλλη μια φορά εκπρέσωμαι για το γεγονός ότι οι εκβιασμοί της μαροκινής κυβέρνησης έφεραν αποτελέσματα για πολλούς συναδέλφους μες στο σώμα αυτό. Δεν ήταν εδώ ψηφοφορία για υπέρ ή όχι μιας κυβέρνησης, αλλά κατά πόσο συνάδει με το διεθνές δίκαιο ή όχι μια τέτοια συμφωνία. Πρόκειται για μια παράταση της συμφωνίας με το Μαρόκο χωρίς προηγουμένως να έχει δώσει την ε, γνωμοδότησή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό έκανε η Επιτροπή. Η τωρινή συμφωνία επιτρέπει σε δικά μας σκάφη να πηγαίνουν στη Δυτική Σαχάρα, στα δικά της ε, δηλαδή ύδατα, χωρίς ε, εκείνοι να έχουν δώσει την γνώμη τους. Είναι παράνομο αυτό πρέπει αν μη τι άλλο να δεχτείτε ότι υπάρχει μια αβεβαιότητα. Γι' αυτό και εμείς θεωρήσαμε ότι έπρεπε να πάει υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να γνωμοδοτήσει και να μας βοηθήσει να πάρουμε μια σωστή απόφαση για ένα θέμα το οποίο έχει και πολιτικές αλλά και οικονομικές και οικολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Λυπούμε λοιπόν που περισσότεροι συνάδελφοι δεν το κατάλαβαν με τον ίδιο αυτό τρόπο και με την αρνητική τους ψήφο οδηγούν σε μια κατάσταση άδικη και νομικά απαράδεκτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν να τελειώσουμε, έχω μια ανακοίνωση. Από την ομάδα των φιλελεύθερων μου έχει ζητηθεί να ορίσω τον Γιβένε Μαρίνη όσον να αντικαταστήσει τον ε, Τζαμάρο Ούγκιας που ήταν στην Επιτροπή Μεταφορών και αντικαθιστά τον Βιτσέντσο Γιοβίνε. Υποθέτω ότι εγκρίνεται, αφού δεν βλέπω καμία αντίρρηση.